Κυρίε και κύριοι, σας ε, παρακαλώ να αρχίσουμε. Θέλω να σας χαιρετήσω εγκάρια. Θα αρχίσουμε σήμερα. Με την τροποποιημένη μερσία διάταξη. Δηλαδή για το διάστημα θέλουμε να υποβάλουμε λεπτομερείς ε, ερωτήσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή και από την ευκαιρία της έκθεσης REMIC είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και είδαμε ότι υπήρχαν πολλά ανοιχτά ερωτήματα που θέλαμε να διευκρινίσουμε. Υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον της Επιτροπής εδώ. <laughs> Αλλά τώρα βέβαια είμαστε πολύ ολιγάριθμοι. Είναι παρούσα η Εκτελεστική Επιτροπή. Ορισμένοι συνάδελφοι υπέβαλαν γραπτέ ερωτήσει και μπόρεσε να προετοιμαστεί η Κομισιόν. Και περί αυτού επρόκειτο ότι δεν θέλαμε να γενικολογούμε, αλλά να εξετάσουμε συγκεκριμένα σημεία. Η πρότασή μου είναι, αν συμφωνείτε συνάδελφοι, να δώσουμε καταρχήν το λόγο στην Επιτροπή για να μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις που υποβάλλουμε και μετά ίσως να συζητήσουμε. Μου φαίνεται ότι θα ήταν το πιο συνετό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συνετά. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φέρχοφ, παρακαλώντα τον να αναφερθεί στα ερωτήματα που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι. Έχετε νομίζω τις ερωτήσεις. Εντάξει, ωραία. Κύριε Φέρχοφ. Καλημέρα σας. Και σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ίσως σαν γενική εισαγωγή θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πριν περάσω στις συγκεκριμένε ερωτήσεις. Και μετά θα περάσω στις ε, λεπτομέρειες. Καταρχήν είναι σημαντικό να θεωρήσουμε πού βρισκόμαστε και τι σημαίνει το Γαλιλαίο. Το Γαλιλαίο είναι θέμα υποδομών. Αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από μερικά χρόνια. Είναι σαφές για όλους. ότι η Ένωση προσφέρει προστιθέμενη αξία για τα προγράμματα αυτά, μια που είναι πάρα πολύ ακριβά για ένα ομονωμένο κράτος. Οι υποδομές ε, ε, συμβάλλουν στην ε, βασική λειτουργία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την στρατηγική του 2020, όσον αφορά τις καινοτομίες και πιο πράσινη και συνδεδεμένη ανάπτυξη και οικονομία, καλύπτουν και άλλους στόχους. Μέχρι στιγμή η συνολική επένδυση του Δημοσίου Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,4 δις ευρώ περίπου από το 2000 έως το 2013. Δέκα έτη μελέτης αναπτύξης τεχνολογίας, ε, πρόθεσης πληρολογίας, δημιουργία γνώσεων, βιομηχανικές αναπτύξεις, ε, διεθνείς συμφωνίες, ε, διεθνείς διεθνές και πλήρε πλαίσιο για τη διακυβέρνηση, όλα αυτά τα έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα συστήματα αυτά κοστίζουν πολύ χρόνο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ε, θα υπάρξουν νέα συστήματα στις αεροπορικές μεταφορές, ιδίως όσον αφορά την ασφαλεία της ζωής. Ε, ε προβλέπει δορυφόρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται για να εκτοξευθούν του χρόνου. Η πρώτη εκδόση θα γίνει το επόμενο έτος και θα ήθελα να σας πω πάλι ότι ε, και εδώ έχουμε εργαστεί πάρα πολύ. Θα πρέπει να εξετάσουμε τώρα μακροπρόθεσμα. Η χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση για το Καλλιό και το ΕΚΝΟΣ δεν είναι επιδοτήσεις για υπηρεσίες, αλλά επενδύσεις ε, πραγματικές. Και οι μελλοντικέ ε, προκλήσεις ποιες είναι. Για το έκνος χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την, ε, τις υπηρεσίες του Γαλιλαίου στις αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, γεωργία κλπ. για να μειώσουμε το χρόνο επενδύσεων, βελτίωση των κυκλοφορικών συστημάτων, ανάλογα και στους ε, ναυτιλιακούς και άλλους τομείς. Ε, για το Γαλιλαίο έχουμε δύο φάσεις μπροστά μας. Πρώτον, πώς θα προχωρήσουμε με την αρχική ιδέα και τι χρειάζεται για τις κατόπιν λειτουργίες και εφαρμογή μακροπρόθεσμα. Η πρώτη φάση, αυτό το λεγόμενο ramp-up, είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουμε. Αν θα, έχουμε γλίγορη και όχι τόσο ακριβή προσέγγιση ή μια πιο αργή και ε, πιο ε, ακριβή. Ε, αν έχουμε την πιο γλίγορη και λιγότερο ακριβή, χρειαζόμαστε συμπληρωματική χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φύση, στη λειτουργική φύση, μετά την πλήρη εγκατάσταση των ε, απαραίτητων μηχανισμών, θα πρέπει να φροντίσουμε οι χρήστες να επενδύουν στο υλικό που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Θα πρέπει να πούμε ότι οι εταιρείε όπως η Air France, η KLM ή η Lufthansa δεν θα επενδύσουν σε υλικό ή σε εγκρίσεις ή καν σε με εκπαίδευση, εάν δεν έχουν εμπιστοσύνη στη λειτουργία του συστήματος για μια μακρά περίοδο δεκαετιών. <coughs> το Καλλιλέο απαιτεί 27 δορυφόρους σε πλήρη λειτουργία ε, κάθε στιγμή, άσχετα αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ε, κακές λειτουργίες κλπ. χρειαζόταν οπωσδήποτε 27 δορυφόροι. Και όλοι οι συλλομπραντικοί δορυφόροι που εκτοξεύονται χρησιμεύουν για να καλυφθούν ενδεχομένα προβλήματα στους 27 βασικούς. Αυτή τη στιγμή, και απαντώ ήδη σε μια ερώτηση, έχουμε προχωρήσει με 18 δορυφόρους. η οποία θα λειτουργεί κατά 95% του χρόνου. Γιατί τρεις, αυτό σημαίνει ότι τρεις εβδομάδες το χρόνο αυτοί οι δορυφόροι δεν θα σας δίνουν καμία δυνατότητα να δείτε πού βρισκόσαστε. Λοιπόν υπάρχουν όμως πάρα πολλοί χρήστες που απαιτούν πλήρη ε, ενημέρωση του στίγματός τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Περιμένουν λοιπόν να υπάρχουν και οι υπόλοιποι χρειάζονται για μεταφορές, για τις αποστολές ειρηνευτικού τύπου, για διάφορες ε, κυβερνητικέ ε, αποστολές κλπ. κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζονται συμπληρωματικές επενδύσεις για να μπορούσε ε, αυτό το υλικό να διατηρηθεί σε κατάσταση λειτουργίας σε γενικές ε, γραμμές το Γαλιλαίο και οι έγκμες είναι η ακρογωνία λύση των υπηρεσιών που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες και σε όλο τον κόσμο. Προχωράμε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να δούμε μακρυπρόθεσμα τι γίνεται. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να αναφερθώ τώρα σε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί. 14 έχω, αν δεν κάνω λάθος. Και θα τις απαντήσω αν θέλετε μία-μία. Αν θέλετε να μειώσετε το χρόνο ομιλία μου να μου το πείτε. Πρώτη, πόσο εξαρτάται η, θέση, η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τους δορυφόρους αυτούς ε, για την εξέβριση του στίγματος και έχετε σκεφτεί θέματα όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κατερχήν, η αγορά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται για το 2010 17 δις. 17 δις. Αυτό σημαίνει έσοδα από εταιρείε που είναι άμεσα εμπλεκμένες στην πλοήγηση με δορυφόρους, στους εκείνους που αναπτύσσουν ε, το λογισμικό κλπ. κλπ. Η GNSS αφορά πολύ στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Η μελέτη που αξιολογεί το ρόλο που παίζουν τα μηνύματα GPS στην οικονομία αποδεικνύουν ότι πολλές όπως οι τηλεπικοινωνίες εξαρτώνται απόλυτα από το GPS. Αυτά τα μηνύματα έχουν σαν στόχο να συγχρονιστούν τα διάφορα δίκαια και αν δεν συγχρονιστούν πάβουν να λειτουργούν. η, η, απο, απώλεια από τη μη λειτουργία είναι της τάξης του 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα. Έχει γίνει μια ανάλυση κοστος ωφελίας και θα βρείτε πολλά στοιχεία για τη σημασία της πλοήγησης με δολοφόρους για την οικονομία εκεί. Σε σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θα σας κάνω μια απλή παρουσίαση. Είναι πολύ υψηλότερη η απόδοση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης. Το εσωτερικό ποσοστό επιστροφής του γολίου είναι της τάξης 40%, ενώ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι μόνο 7 έως 8%. Δεύτερο ερώτημα η Κομισιόν εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη για πιο ε, μη στρατιωτική ε, χρήση του Γαλιλαίου ή χρησιμοποιείται κυρίως για τις ειρηνευτικές αποστολές. Θα ήθελα να σας πω ότι βέβαια η απόφαση του γιατί θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό είναι μια απόφαση που λαμβάνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από κοινού. Αυτή τη στιγμή θεωρείται μη στρατιωτικό και υποπολιτική υποπολιτικό έλεγχο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν σίγουρα τομείς όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι δυνατή και η χρήση στρατιωτικού τύπου, παραδείγματο χάρη για την μεταφορά των στρατών, γιατί θα πρέπει να υπάρχει εκεί πρόβλημα. Οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι είναι στρατιωτική χρήση και τι δεν είναι εάν κανένας εξετάσει τον νομικό καθεστώς ορισμένων μονάδων. Η συζήτηση λοιπόν άλλων χρήσεων είναι ακόμα ανοιχτή, όπως σας είπα. Αλλά νομίζουμε ότι αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση που θα πρέπει να γίνει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και η Κομισιόν θα εφαρμόσει απλώς την απόφαση που θα ληφθεί. Σύντομα, η Κομισιόν θα σε υποβάλει μια πρόταση για τη χρήση του μηνύματος PRS που αφορά ε, καταρχήν μια συζήτηση για το πού θα χρησιμοποιείται αυτό και πώς θα οργανωθούμε. Επίσης, ε, κάναμε κάποιες έρευνες στα κράτη-μέλη για να δούμε πόσο ενδιαφέρονται για τη χρήση του PRS και υπάρχουν πάρα πολλέ κυβερνητικέ υπηρεσίες που ενδιαφέρονται στα κράτη-μέλη, παραδείγματος κανονισμένοι τομεί Άμυνα μέχρι την προστασία των πολιτών και πολλά άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε θα πρέπει το σύστημα να προστατεύεται σωστά, είναι μια πολύ κρίσιμη υποδομή. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα ασφάλειας επίσης και γι' αυτό θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να το προστατεύσουμε αυτό το σύστημα. είναι το ερώτημα που μας υποβάλλατε. Πώς αξιολογεί η Κομισιόν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής εργάζονται στην τρίτη γενιά του GPS, η Ρωσία ολοκληρώνει το σύστημά της και η Κίνα έχει ξεπεράσει την Ευρώπη στην δημιουργία του δικού του συστήματος. Τι θα κάνει η Ευρώπη για να είναι πλήρως ανταγωνιστική και κυρίαρχη σε αυτό το τομέα. Είναι σωστό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Ε, αυτή τη στιγμή εκτοξεύουν τους λεγόμενους 2F δορυφόρους, 2F satellites. Και από το χρόνο θα ξεκινήσουμε το GPS 3. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε. Υπάρχουν πάντα ονομαστικοί χρόνοι που δεν τηρούνται, καθυστερήσει κλπ. Θα πρέπει να δούμε τελικά ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, είναι χρήσιμο να πούμε ότι οι συζητήσεις στην Ευρώπη για τον Καλλιλέο προώθησαν τη ΣΥΠΑ αλλά και την Κίνα, τη Ρωσία και την Ιδία να εξετάσουν τα δικά τους συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Η δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους έκανα τις άλλες να κατανοήσουν καταρχήν ότι τα συστήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, κατά δεύτερον οι μη στρατιωτικές χρήσεις είναι επίσης όσο πάει και πιο σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη, εάν εμείς θέλουμε να δώσουμε στο Γαλιλαίο και στο ΕΓΜΕΣ τη δυνατότητα να μας προσφέρουν αυτές τις ε, υπηρεσίες, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα παράθυρα ευκαιρίες που μας αφήνουν τα άλλα συστήματα. Αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε το Γαλιλαίο να είναι το δεύτερο σύστημα επιλογής όπως το αποκαλούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να θεωρήσουμε ότι θα πρόκειται να είναι εύκολο ή δυνατό να ξεπεράσουμε το GPS, να το αφήσουμε κατά μέρος. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά παρόλα αυτά είναι καλό να έχουμε ένα δεύτερο σύστημα επιλογής. Εργαστήκαμε αρκετά για να προωθήσουμε αυτή την ιδέα, ιδίως συμφωνείς με τη ΣΥΠΑ, για να πετύχουμε την εμπιστοσύνη της ε, Αμερικανικής βιομηχανίας ότι το Γαλιλαίο είναι σύστημα που μπορούν να επιλέξουν αντί του GPS ή εκτός του GPS. Το ρωσικό σύστημα αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Και βέβαια έχουμε και το σύστημα των Κινέζων, όπου δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο έχουν προχωρήσει. Νομίζω ότι προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα προς το εμπρός, αλλά υπάρχουν πολύ αντιφατικές πληροφορίες σχετικά. Τούτον ενώ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να έχουμε ένα πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας και να τοποθετήσουμε σωστά τον Γαλιλαίο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με τον Γαλιλαίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τέταρτη ερώτηση με τη νέα βελτίωση του GPS που προβλέπεται για το 2014 και 2018 και την νέα κινητική τεχνολογία υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που προσφέρει το Γαλιλαίο και να παραμείνουμε ενδιαφέροντες και ελκυστικοί για τους ανταγωνιστές μας. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν προβλέψει οι άλλες, τα άλλα συστήματα, ιδίως εμπορικές ε, υπηρεσίες και οι η υπηρεσία PRS που είναι διαφορετική από την απλή ε, χρήση. Και επίσης έχουμε κάτι που δεν έχουν σκεφτεί καθόλου τα άλλα συστήματα, δηλαδή αναζήτηση και διάσωση. Τρεις από τις πέντε υπηρεσίες λοιπόν που προσφέρουμε είναι διαφοροποιημένες από το υπόλοιπο. Πήραμε μία γνώση μας απόφαση ότι οι ανοιχτές υπηρεσίε αυτές θα είναι συμβατές με το GPS και έχουμε τις απαραίτητες συμφωνίες στα χέρια μας για να το πραγματοποιήσουμε. Τώρα το πώς οι δορυφόροι θα υπάρξουν αυτό εξαρτάται από τους πόρους που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Θα είναι επαρκές το σύστημα για να είναι ανεξάρτητο. Τα νούμερα τώρα. Έχουμε ήδη αναθέσει συμβάσεις για τρία πακέτα έργου εκτό από τα έξι, τρία, τρεις δέσμες έργων, το System Support Contract 85 εκατομμύρια για 14 δορυφόρους 560 εκατομμύρια και προβλέπουμε 5 πυράβλους Soyuz και 390 εκατομμύρια, δηλαδή τη χρήση των πυράβλων αυτών, 390 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, οι πόροι που δεν έχουν ακόμα διατεθεί αναφέρονται σε ε, εκτοξεύσεις που θα γίνουν ακόμη και τα πακέτα έργων για τον τομέα αποστολών και επιχειρήσεων και αναμένουμε οι συμβάσεις αυτές να αρχίσουν να εκπονούνται μετά το καλοκαίρι. Με τον προπολογισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε εν τέλει να εκτοξεύσουμε 18 δορυφόρους, τους 14 που είναι έτοιμοι και άλλους 4 και έχουμε και αυτό που προβλέπουμε ως αρχική επιχειρησιακή ικανότητα που θα προβλέπει μια ανοιχτή υπηρεσία PRS και αναζήτηση και διάσωση. Έχουμε επίσης και την αναζήτηση και διάσωση, όπως είπα, για τη διάσωση ζωής, η οποία ε, δεν θα είναι, οποίες δεν θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, αλλά 95%. Δηλαδή για τρεις εβδομάδες τον χρόνο συνολικά δεν θα είναι διαθέσιμες αυτές οι υπηρεσίες, διότι δεν υπάρχουν απαρκείς δορυφόροι. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι ο Γαλιλαίος είναι σύστημα 27 δορυφόρων μαζί με την χερσαία υποδομή ελέγχου. Δεν είναι δηλαδή ένα πλήθος δορυφόρων όπου καθένας κάνει τα δικά του. Κάθε δορυφόρος συμβάλλει στη λειτουργία του συνολικού συστήματος. Άρα χρειαζόμαστε το όλο σύστημα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και για να λειτουργήσει το σύστημα. Αν μου επιτρέπετε την σύγκριση, είναι κάπως σαν να πάτε να, να παραγγείλετε ένα αυτοκίνητο. Δεν τίθεται θέμα ότι θα έχει τέσσερις τροχούς. Έτσι λοιπόν και ο Γαλιλαίος βασίζεται σε έναν αριθμό 27 δορυφόρων και τους χρειαζόμαστε για τους 27. Δεν είναι το θέμα πόσες ρεζέρβες θα χρειαζόμαστε στο αυτοκίνητο. Πάντως, εμείς για την ώρα θεωρούμε ότι θα υπάρχουν τρεις δορυφόροι εφεδρικοί, άρα συνολικά θα φτάσουμε στους 30, αλλά ακόμα το μελετούμε. Πρέπει να φτάσουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα. Οι χρήστες στις αγορές περιμένουν την ικανότητα αυτή για να προχωρήσουν και αυτοί σε επενδύσεις από την πλευρά τους, ως χρηστών δηλαδή. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί που έχουμε δηλαδή μπροστά μας αυτή τη στιγμή για την ολοκλήρωση του συστήματος. Και γι' αυτό έχουμε καθορίσει ε, κάποιες, κάποια ενδιάμεσα στάδια και ε, μελετούμε και την τελική χρηματοδότηση. Τώρα, η μετρίαση των κινδύνων που ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποια μέτρα λαμβάνονται, μας ρωτάτε. Και επίσης αν έχουν ε, ληφθεί υπόψη οι κίνδυνοι της ηλιακής ακτινοβολίας. Τώρα πρώτα για την μετρίαση των κινδύνων. Έχουμε εντάξει στο σύστημα μια λειτουργία Διαχείριση του κινδύνου. Είναι σημαντικό όταν αναπτύσσεται ένα τέτοιο σύστημα να κατανοούνται οι κίνδυνοι. Εάν κανεί παραμείνει μονάχα σε μια συζήτηση του κόστου, αυτό μπορεί να αποκρύψει το γεγονό ότι πίσω από το κόστο μπορεί να κρύβονται κίνδυνοι οι οποίοι αν υλοποιηθούν οδηγούν σε απότομη αύξηση του κόστους. Λοιπόν, εγώ θα ζητούσα από όλες και όλους οι οποίοι εξετάζουν το θέμα αυτό να εξετάσουν το θέμα και από την πλευρά του κόστους και από την πλευρά των κινδύνων. Πάντοτε θα υπάρχουν κίνδυνοι διακοπής της λειτουργίας διακοπής της λειτουργίας της τεχνολογίας ε, πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, ήδη έχουμε μια καθυστέρηση στην παράδοση των ε, δορυφόρων IFE, διότι υπάρχει ένα ε, τμήμα τους ένα κουτί, το οποίο δεν λειτουργεί. Και μιλούμε τώρα για προβληματική λειτουργία ενός μονάχα τμήματος του συστήματος που δεν λειτουργεί. Έχουμε λοιπόν μελετούμε τους ε, ε, κινδύνους, μετρίαση των κινδύνων, συζητούμε με την ε, European Space Agency, Έχουμε risk management σε όλα τα επίπεδα των ε, προμηθειών, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κύριε Φερχόφ, αρχίζουμε και αντιμετωπίζουμε πίεση χρόνου. Μπορείτε να τα πείτε κάπως πιο ε, γρήγορα, γιατί και μη λησμονείτε ότι 10 η ώρα έχουμε ψηφοφορίες. Αν Χαίρομαι για τις πλήρες απαντήσεις σας. Αν όμως οι συνάδελφοί μου θέλουν να ρωτήσουν, να θέσουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, ε, δεν θα έχουμε πια τον χρόνο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έρχομαι στο επόμενο θέμα. Ε, σχετικά με το double sourcing, τις διπλές πηγές δηλαδή δορυφόρων που είναι μετρία του κινδύνου, δηλαδή αν θα έχουμε εφεδρικές πηγές, για παράδειγμα και για την ε, προμήθεια των δορυφόρων και για τις εκτοξεύσεις, ώστε εάν μία από αυτές δεν λειτουργήσει, μία από αυτές τις πηγές δεν λειτουργήσει, να έχουμε μία άλλη. Βέβαια αυτές οι εφεδρικές πηγές, το double sourcing αυτό, ε, σημαίνει έξτρα κόστος. Εάν όμως υλοποιηθεί κάποιος κίνδυνος θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα ιδιαίτερα για τους δορυφόρους και επίσης για τα συστήματα εκτοξεύσεως. Αυτά είναι κρίσιμα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ώστε το σύστημα πλογήσεως, το ευρωπαϊκό σύστημα Πλογήσεως, ένα λεπτό να διαβάσω πιο κάτω, των 30 δορυφόρων θα μπορεί να λειτουργήσει και να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που προβλέπονται. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε πρόσθετη χρηματοδότηση και γίνονται σε υψηλότερο επίπεδο μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη συζητήσεις για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η έξτρα χρηματοδότηση. Και αν είναι λογικό ήδη τώρα να ε, υποβληθούν οι αιτήσει για την έξτρα χρηματοδότηση ή αν θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη περίοδο. Η επόμενη ερώτηση ποιες είναι οι ημερομηνίε για τη λήξη της χρηματοδότησης προμήθεια των ε, ε, δορυφόρων στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική και ούτω καθεξής. Εάν δεν γίνουν αυτά μέσα στο 2012, τότε θα έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις και τουλάχιστον τριετή καθυστέρηση στην πλήρη επιχειρησιακή ε, λειτουργία, πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε παράθυρα ευκαιρίας εάν δεν το κάνουμε. Επίσης θα αυξηθεί το κόστος, γιατί θα χρειαστεί να κόψουμε τις προμήθειες σε μικρά κομμάτια και θα έχουμε επομένως σημαντική αύξηση του κόστους. Επίσης κάθε κενό στην παραγωγή σημαίνει ότι οι βιομηχανίες που παράγουν τα ε, διάφορα, τα διάφορα μέρη του συστήματος δεν θα μπορούν να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό που ε, εργάζεται σε αυτές και επομένω θα χαθεί μια συνέχεια. Όπως είπα λοιπόν, η παρούσα χρηματοδότηση συζητείται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή και ελπίζουμε στις επόμενες εβδομάδες να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το εάν θα ζητήσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση. Πάντως είναι ε, σαφής οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων. Το χρονοδιάγραμμα τώρα για την εκτόξευση των δορυφόρων. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Προβλέπονται για τα μέσα του 2011 και για το τέλος του 2011. Πρόκειται για καθυστέρηση, όπως είπα, γιατί οφείλεται σε, στην αδυναμία λειτουργίας ενός τμήματος του δορυφόρου, ενός κουτιού του δορυφόρου, των δορυφόρων οι συμβάσεις για τους 14 πρώτους FOC δορυφόρους προβλέπεται να αρχίσει η εκτόξευσή τους από το τέλος του 2012 στη διάρκεια του 2013 και στις αρχές του 2014. Αν όλα, αν όλα λοιπόν πάνε καλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντοτε σε διαστημικά προγράμματα πάντως αυτό που προβλέπεται είναι και οι 18 δορυφόροι να βρίσκονται στο διάστημα στο πρώτο εξάμεινο του 2014. Η επόμενη ερώτηση είναι πόσα χρήματα αναμένεται να χρειαστούν στις, στα επόμενα ε, δημοσιονομικά πλαίσια. Οι προβλέψεις που έχουν γίνει για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του συστήματος και του Γαλιλαίου και του Έγνος συν έξα χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούμε κατά μέσον όρο περίπου 750 εκατομμύρια τον χρόνο. για τα επόμενα χρόνια. Με αξίες του 2010 και 2011. Υπάρχουν ορισμένα δημοσιονομικά θέματα που προκύπτουν Γιατί αν θέλουμε να αγοράσουμε το σύστημα όπως κάνουμε συνήθως με δημόσιες προμήθειες, δηλαδή το χαμηλότερο κόστος, θα έπρεπε να έχουμε ε, διαφορετικού είδους ε, προμήθειες σήμαινε δηλαδή διαφορετικές πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών. Αυτό για την ώρα είναι δύσκολο στον προϋπολογισμό θα, χρειαζόταν τότε να κατακαιρματίσουμε τις συμβάσεις σε μικρότερα κομμάτια και το κόστος του συστήματος θα αυξανόταν. Πάντως για τα δύο συστήματα έγνωση και γαλιλαίος 750 εκατομμύρια τον χρόνο για το επόμενο διάστημα. Μόνο το GPS, σας δίνω ένα συγκριτικό στοιχείο, κοστίζει ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Μόνο το GPS. Σας ε, δίνω λοιπόν μια ιδέα του, του κόστους των συστημάτων αυτών. Τρεις ερωτήσεις μου μένουν ακόμα. Ήδη από το 1995 ε, θεωρούσαν οι ΗΠΑ ότι θα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό το GPS. Γιατί δεχθήκατε το επιχείρημα ότι ο Γαλιλαίος μπορεί να είναι εμπορικά βιώσιμος. Θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει ο Γαλιλαίος με επαρκή έσοδα ώστε να είναι αυτόνομος. Οι μελέτες που έχουμε κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο μας δείχνουν ωστόσο ότι αυτή η ιδέα δεν είναι σωστή. Δεν είναι αυτό δυνατό. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια αγορά για τις εμπορικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Γαλιλαίος που θα αποδίδουν 50 με 70 εκατομμύρια τον χρόνο όταν θα έχει οριμάσει η αγορά αυτή και ίσως υπάρχει και μια αγορά για το PRS. Για το PRS υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όπου δηλαδή ναι μεν τα Υπουργεία Οικονομικών και τα Υπουργεία Μεταφορών θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι επιπληρωμή τα ε, Υπουργεία όμως τα οποία ε, θα κάνουν χρήση του συστήματος αυτού, τα Υπουργεία χρήστες, θεωρούν ότι το σύστημα έχει ήδη πληρωθεί από χρήματα του δημοσίου και άρα δεν πρόκειται να πληρώνουν τίποτα. Η μόνη υπηρεσία από την οποία μπορούμε να αναμένουμε έσοδα είναι η εμπορική υπηρεσία και όπως είπα 50 με 70 εκατομμύρια κατά μέσον όρο του χρόνου και βεβαίως εν ώψη του κόστου του συστήματος δεν υπάρχει θέμα να είναι ε, βιώσιμο, αυτόνομα το σύστημα. Από αυτό προκύπτουν ορισμένε επιπτώσει, ότι δηλαδή ο δημόσιο τομέα χρειάζεται να οργανωθεί και από πλευρά διακυβερνήσεω για να ε, χειριστεί το σύστημα. Η ε, πλοήγηση υψηλής, η τεχνολογίας θα ορίζεται από τις ΗΠΑ το Γαλιλαίο θέλει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσει να αδράξει τους καρπούς από αυτό το εγχείρημα. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός αρκεί να ε, εκμεταλλευτούμε τις υποδομές. Να σας δώσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Η ενδυνάμει αγορά για τη δορυφορική πλοήγηση και υπηρεσίες ανά τον κόσμο στα επόμενα χρόνια θα ανέρχεται σε 220-240 δις ετησίως. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα ήθελε το 1 τρίτον αυτής της αγοράς, δηλαδή 70 δις ευρώ ετησίως. Αυτός θα ήταν ο στόχος της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτό είναι το επιθυμητό. Καταρχήν θα πρέπει να επενδύσουμε στο δικό μας σύστημα δηλαδή 750 δις ετησίως, 750 ε, εκατομμύρια ετησίως με συγχωρείτε και το υπόλοιπο θα ήταν για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη από την European Space Agency και από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Έχουν γίνει συγκρίσεις και ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία στις ΕΠΑ. Το ομοσπονδιακό πρόγραμμα είναι της τάξης των 200 με 500 εκατομμυρίων ετησίως. Άρα, εάν μιλάμε για πολιτική χρήση, όχι στρατιωτική χρήση δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε κάτι το αντίστοιχο μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα σε αυτό το τομέα. Τελευταία ερώτηση. Πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τη συνεργασία με την Κίνα. Ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι διακοπής λειτουργίας. Πώς αυτό θα πλήξει το πρόγραμμα ασφάλειας Ευρώπης και διαχείρισης του Γαλιλαίου. Η κατάσταση με τους Κινέζους εταίρους είναι αρκετά περίπλοκοι. Αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την συμβατότητα συχνότητας και αυτό αφορά και τις σχέσεις τους με τις ΕΠΑ. Και είπα και εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύσεις γι' αυτό. Ε, γίνονται πολυμερείς και διμερείς συζητήσεις επί του θέματος. Θα έχουμε μία πολυμερή διαβούλευση τον Οκτώβριο και από όσο γνωρίζω ήδη και την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, στα Ηνωμένα Έθνη και τον ε, Ιούλιο θα έχουμε διμερείς σχέσεις με την Κίνα. Ελπίζουμε να εξευρεθούν λύσεις. Εάν δεν προβλεφθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το λειτουργικό του Γκαλιλαίου για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Νομίζουμε ότι αυτό είναι κατόρθωτο και είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν τρόποι διεξόδου. Το ιδεώδες θα ήταν να γίνουν συζητήσεις με την Κίνα και ενδεχόμενη συμφωνία. Μετά από την επιστολή του Πρόεδρου Μπαρόζο και την απάντηση των, Κίνες, αρχών της Κίνας, ε, έχουμε σοβαρές ελπίδες για κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και ήταν όντω σημαντικό να απαντηθούν. Αλλά όπως είπα 10 η ώρα έχουμε ψηφοφορία. Ο κ. Οντί. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, μακροσκελέστατες απαντήσεις. Θα ήθελα να επαναλάβω ενώπιον του υπευθύνου της Κομισιόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει σε πολλά θέματα και το πρόγραμμα Γαλιλαίο ε, ανελήφθη από την Κομισιόν υπό τον Επίτροπο Μπαγό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις επεξηγήσεις. Θα πρέπει η Επιτροπή να μας εγγυηθεί ότι θα επιτύχουμε διαφορετικά θα έχουμε εκ νέου μία αποτυχία. Η ερώτησή μου τώρα. Θεωρούμε ότι το Γκαλιλαίο είναι το αντίπαλο δέος του GPS. Τη στιγμή που θα υπάρχει παγκόσμια διακυβέρνηση G20 κλπ. Αντί να είμαστε ανταγωνιστικοί δεν θα πρέπει να είμαστε συμπληρωματικοί ως προς τους Αμερικανούς ε, και ως προς το GPS για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα με τους φίλους μας τους Αμερικανούς. Να μην είμαστε δηλαδή σε σχέση ανταγωνισμού. Γεια Χολ. Ευχαριστώ Επιτροπή. Πολύ ενδιαφέρουσες και πλήρης απαντήσεις. Δύο πράγματα δεν απαντήθηκαν που περιλαμβάνονταν μεταξύ των ερωτήσεων. Ποια είναι η κατάσταση από τις ε, ιδιακές εκρήξεις και δεύτερον είναι αλήθεια ότι ο πρόσθετος προϋπολογισμός θα είναι της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων ή ευρώ μάλλον, συγγνώμη. Και σε προηγούμενη συζήτηση με την Επιτροπή υπονοήθηκε ότι οι δυσκολίες με την Κίνα είναι ότι η κυβέρνηση και ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός δεν κινούνται απολύτως εκ παραλίλου και ότι το πρόβλημα θα ήταν στην πραγματικότητα ο Κινέζικο στρατό, ανεξαρτήτω του τι λέει η κυβέρνησή τους. Ευχαριστώ Λάμπερτ. Θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο Ζαμπιέρο Το να ζητήσουμε εγγύηση από την Κομισιόν είναι σαν να τη ζητάμε κάτι το οποίο δεν, μπορεί να κάνει. Όχι ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Και Μιλάμε για ε, αρκετά κονδύλια. Αν δεν μπορούμε να διαθέσουμε 750 εκατομμύρια ετησίως, τότε το σύστημα δεν θα είναι λειτουργικό. Σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους γιατί αντιμετωπίζουμε όχι μόνο αυτό το project αλλά ε, και στο πρόγραμμα ITER έχουμε υπερβεί τον προϋπολογισμό μας. Ή δηλαδή, είτε δηλαδή θα δεχτούμε τα δεδομένα όσα έχουν και θα αγοράσουμε ολόκληρο το σύστημα, διαφορετικά ας το αφήσουμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι το ζήτημα κατά πόσο διαθέτουμε τα κονδύλια, αλλά μπορούμε να το κάνουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό το σύστημα όχι μόνο για 5 ή 10 χρόνια, αλλά μακροχρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία επιτάπητος για να λάβουμε αυτή την απόφαση και νομίζω ότι δεν διαθέτουμε όλα τα στοιχεία. Είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να προωθηθεί με το Συμβούλιο κάποια στιγμή, γιατί βρισκόμαστε, βρισκόμαστε και δεν μπορούμε να αρκεστούμε στα αρχικά δεδομένα ικανότητας. Αν προχωρήσουμε, αυτό θα έχει επιπτώσεις, δηλαδή θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα αποκλείσουμε κάτι άλλο. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν είμαι σίγουρος ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Κύριε Νίμπλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, Ευχαριστώ βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί πραγματικά εξαιρετικό έργο. Κύριε Φερχόφ, χαίρετε τη απολύτω εμπιστοσύνη μου. Και κάτι τέτοιο δεν το λέω συχνά στην Επιτροπή. Δεύτερο, επί τη ουσία. Συμφωνώ με του δύο προηγουμένου, Οντί και Λάμπερτ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπή. Και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώ θέλουμε. Εάν θέλουμε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, τότε πρέπει να φροντίσουμε να εξασφαλιστούν όλες οι πολιτικές προϋποθέσεις, ώστε το σύστημα αυτό να καταστεί λειτουργικό το δυνατόν συντομότερο και να μπορέσει να λειτουργήσει εμπορικά. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να είναι σαφή τα κοστολόγια. Εάν αυξάνουν τα κοστολόγια, αν αυξάνει το κόστος, πρέπει να το ξέρουμε από τώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συνολική επισκόπηση του κόστους και τότε θα κληθούμε να λάβουμε την απόφαση. Ακούστηκε προηγουμένω μια παρατήρηση για το ίτερ, το οποίο είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξή μα. Εάν δεχθώ ε, τα όσα λένε οι εφημερίδε, φαίνεται από τα 2,4 δι ευρώ το κόστο του να έχει ανέρθει στα 7 δι ευρώ. Χρειάζεται λοιπόν και εκεί και εδώ να λάβουμε ξεκάθαρε αποφάσει για το πού θέλουμε να βαδίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ισοδύναμη και ισότιμη και παγκοσμίω. Ο κύριος Έλερ. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Νίμπλερ και με τον κύριο Λάμπερτς. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου η mid-term review ερμηνεύεται από την κοινή γνώμη ως το ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο, στη δημοσιονομική προοπτική 8, ενώ ακόμα δεν έχουμε βγει από την 7. Από όσο γνωρίζω από τα ποσά του προϋπολογισμού, δεν είναι καλυμμένα τα πράγματα αυτά από τον προϋπολογισμό και διαπραγματευόμαστε νούμερα τώρα τα οποία δεν υπάρχουν ούτε το δημοσιονομικό πλαίσιο 7, ούτε και ε, στο, στο ειδικότερο τμήμα του διαστήματος. Άρα δεν χρειαζόμαστε μια απλή επανεξέταση, review, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα νούμερα. Πριν από το καλοκαίρι συνέρχεται το ε, Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕΡ και πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει mid-term review χωρίς να τα γνωρίζει τα νούμερα αυτά ακριβώς. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βερχόφ, σας διαθέτω τέσσερα λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα υποβάλω, θα ομαδοποιήσω μάλλον τις ε, ερωτήσεις ως προς τη χρηματοδότηση. Να είμαστε απόλυτα σαφείς για τα αίτια του ενδεχόμενου αιτήματο επιπρόσθετη χρηματοδότησης γιατί το Διευθυντήριο δεν έχει λάβει απόφαση στην Κομισιόν και ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να αποφασίσουμε ή πριν το καλοκαίρι. Θα έχουμε όλα τα στοιχεία επιτάπητος. Ξεφύγαμε από το αρχικό ε, κόστος Υπερβήκαμε δηλαδή κατά 600 εκατομμύρια το κόστος και τα κράτη-μέλη ζήτησαν την επιπρόσθετη χρηματοδότηση από εμά διότι δεν μπορούσαν να τα αναλάβουν ε, εκείνα για το δορυφορικό πρόγραμμα. Το δεχτήκαμε γιατί δεν θα μπορούσε να συμπληρωθεί το IAV. Θα έπρεπε να σταματήσει το πρόγραμμα αν δεν γινόταν η επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Μιλάμε για 600 ε, εκατομμύρια υπέρβαση δηλαδή. Το επόμενο θέμα είναι ένα σοβαρό θέμα για τους εκτοξευτές που δεν ελέγχουμε. Είχαμε εκτιμήσεις με την Ευρωπαϊκή Δορυφορική ε, Υπηρεσία σε σχέση με το κόστος το 2007. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί μας το κόστος των εκτοξευτών από το 2000 και μετά κατά 80%. Άρα μιλάμε για 600 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τους εκτοξευτές. Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να αντλήσει από κάπου αλλού ή να φτάσει σε χαμηλότερου κόστους εκτοξευτές. Αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα διότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας και δεύτερον έχουμε το δικό μας πρόγραμμα εκτοξεύσεων και τις δικές μας επιχειρήσεις και έχουμε και δεσμεύσεις δυνάμει του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Έχουμε μία σύμβαση με την Αριάνε Σπάς και εκεί σταματάμε. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε δηλαδή. Άρα μόνο αυτά τα δύο ζητήματα ανέρχονται σε 1,2 δις. Άρα είναι ανεξέλεγκτα πλέον, είναι εκτός ελέγχου μας. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η ιδεατά θα θέλαμε μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση 1,5. Το 1,2 που προανέφερα συν ε, ορισμένα νέα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που σταμάτησαν τη στιγμή που αποφασίστηκαν τα 400 εκατομμύρια από το 2007 και μετά, έτσι ώστε ε, να καλύψουμε τα 3,4 δις που είχαμε ορίσει τότε, μέσα στα πλαίσια και των ε, προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Βλέπετε λοιπόν ότι ως προς τους εκτοξευτές δεν ανέβηκε το κόστος, μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να διαπραγματευτούμε τις τιμές και βρίσκονται, συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις μας δύο χρόνια πριν. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόγραμμα και διαθέτουμε και τα κατάλληλα μέσα. Τεχνολογικά μπορούμε να το κάνουμε, ε, χρησιμοποιούνται οι ε, εκτοξευτές, οι αναθεωρήσεις, μάλλον οι εκθέσεις είναι πάρα πολύ καλές για το δορυφορικό πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε πότε θέλουμε να γίνει πραγματικά λειτουργικό το σύστημα. Και ένα τελευταίο στοιχείο. Μιλάμε για τα δικά μας ε, ε, στοιχεία. Δεν μιλάμε για το ίτερ όπου υπάρχει συνεργασία και ε, με άλλα μέρη του κόσμου. Εδώ κάνουμε επένδυση από τα δικά μας ε, πάγια στοιχεία ενεργητικού στο Γαλιλαίο. Και δεν ζητάμε επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το FP7 ή 8. Δηλαδή δεν μιλάμε για έρευνα και ανάπτυξη πια. Μιλάμε για λειτουργικά έξοδα. Think there uh, Ορισμένες ε, άλλες ε, ερωτήσεις ο κύριος Οντί για τον συνεργασμό με, με την, συνεργασία με το GPS ή τον συμπληρωματικό χαρακτήρα. Το συζητήσαμε με τις ΙΠΑ και βλέπουμε ότι δεν επιθυμούν οι ΙΠΑ ένα κοινό σύστημα με μας. Γιατί, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουμε εμείς, ο πρωταρχικός του στόχος με το GPS είναι στρατιωτικός στόχος και θέλουν να είναι ελεύθεροι να αλλάξουν το σύστημα όπως το επιθυμούν. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή διότι υπάρχει θέμα λήψης GPS στο Αφγανιστάν και αλλάζουν τις συντεταγμένες έτσι ώστε να μπορέσουν να κινηθούν αυτόνομα. Άρα δεν έχουμε ενιαίο σύστημα με το GPS Προσπαθούμε να έχουμε κοινά συστήματα και συμβατότητα καθώς και διαλειτουργικότητα και ένα από τα σκέλη του GPS και του Galileo θα είναι συμπληρωματικά. Σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Χολ για τις ε, ηλιακές εκρήξεις, νομίζω ότι ε, εντάσσονται στα συστήματα IT καινοτομίας και τεχνολογίας δηλαδή. Από ό,τι είδαμε από τις ηλιακές κρίσεις είναι ότι δεν κάνουν παρεμβολές στο σύστημα GPS και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και για τον Γαλιλαίο. Θα το ελέγξουμε δηλαδή. Και η τελευταία απάντηση για το θέμα με τους Κινέζους, τη συνεργασία, είναι γεγονός όπως ε, ξέρετε, ε, το PLA είναι ο βασικός εκτελεστής του προγράμματος. Το θέμα είναι περίπλοκο. Τη στιγμή που υπάρχει ανταπόκριση από τον Πρωθυπουργό της Κίνας, έχουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Αυτές είναι οι απαντήσεις, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Υπήρχαν ούτως ή άλλως και πολλές νέες πληροφορίες και το θέμα του συνολικού κόστους ε, των εκτοξεύσεων μπορεί να μειωθεί ίσως το κόστος ε, αν αναθέσουμε τις εκτοξεύσεις σε άλλους. Αυτό είναι καλό διότι μέχρι τώρα μιλούμε μονάχα για αύξηση του κόστους. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συζήτηση και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Gut. Jo, darf ich äh, die Abstimmung... Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Φαντάζομαι έχετε όλες τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Αν όχι, χάσατε η πρώτη ψηφοφορία για την οργασμό ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Ξέρετε, συνάδελφοι, ότι τον Οκτώβριο 2009 ήδη είχαμε αποφασίσει σχετικά και λόγω της νομική κατάσταση πρέπει να έχουμε εδώ σε απλωστευμένη διαδικασία. Έχετε το χαρτιά μπροστά σας και τα έγγραφα. Καλύτερα αν καθίστε μου φαίνεται, είναι πιο εύκολο να ψηφίσουμε. Λοιπόν, μία ψηφοφορία, νομοθετικό ψήφισμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Ερωτήσεις, Ρόβινς, εντάξει, ωραία, άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. On the left. Λοιπόν, τρεις του ΕΛΚ είναι υπεράριθμοι. Και στους σοσιαλιστές λειτουργούν τα, τα συστήματα. Πολύ ωραία. Τι να κάνω κι εγώ. My God. No? Perhaps you try another one. Για δοκιμάστε το διπλανό. Α, το ίδιο είναι. Όλοι εδώ η αριστερή πλευρά είναι κλειστή. Α.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 για να ξαναδοκιμάσουμε. Κλείνει η ψηφοφορία. Για να δούμε. Okay. Yeah. Okay. Okay. Also, damit... Ωραία. 44. Συνολικά ψηφίσατε. Ναι. Ωραία. Σαν 43 υπέρ. Ωραία. Φτάνει. Πολύ ωραία. Και 46 εδώ δεν λειτουργούσαν. 46-47. Θα προσθέσουμε τους σοσιαλιστές. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Σημαντικό αυτό. Γιατί όλοι στην Ευρώπη θέλουν να ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε εδώ. The next one is um, the Sousa Wagner report. We have there one problem, but I think we can start. Έχουμε τώρα την έκθεση Σόζα Φάκνερ. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 37 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίση 51 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά κατά παρακαλώ αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τριολογικές σκέψεις 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γνωμοδοτήσεις τώρα πολιτιστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κουλτ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κουλτ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 όχι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 22 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται επίση. Τώρα, η χνομοδότηση ΙΜΚΟ. ΙΜΚΟ 1, υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομικές επιτροπές, Ζούρι, 1, 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται επίση. Ζουρί 12 για την 11 υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Ο εστιχής θεωρείται ότι καλύπτεται. Ζουρί 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομοδότηση Νομοδότηση λίπε, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Να ξαναδοκιμάσουμε. Άρχιτε ψηφοφορία. Ein EPP zu viel. Zu three. Τρεις ΕΛΚ υπεράριθμε. Okay. Okay. EPP Τώρα εντάξει. Και οι σοσιαλιστές ακολουθούν να μην έχουν ενέργεια. Α. Closed. Πέρας τα 45 ψηφίσαντες. Θα προσθέσουμε τους σοσιαλιστές. Εντάξει, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Να το ξεχάσουμε. Έκθεση του καλά. Έχετε τα έγγραφα μπροστά σου. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Α, απεσύρθη. Α, συγγνώμη. 22 λοιπόν. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά,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 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. One EPP e too much. Two too much. Δύο και Ωραία. Το πλάσμα σαφές. Και θα προσθέσουμε αυτούς τους οκτώ σοσιαλιστές παρακαλώ. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε την ψηφοφορία. Συγχαρητήρια τους συναδέλφους και συνεχίζουμε με την μερσία μας διάταξη. Έκθεση πρωτοβουλία για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος πλαίσιο. Η συνάδελφος Καβάλιο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, President, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι οι ερευνητές ζητούν εναρμόνιση κανόνων και διαδικασιών και γενική απλοποίηση των κανόνων της υποβολής λογαριασμών. 9.000 ερευνητές υπέγραψαν πρόσφατα αίτηση ζητώντας μεγαλύτερη απλοποίηση στη χρηματοδότηση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν πραγματική ανάγκη αλλαγών και βελτιώσεων στην ε, χρηματοδότηση και στην διοίκηση των προγραμμάτων αυτών. Αποτέλεσμα, ο επίγον χαρακτήρας. Η έκθεσή μας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι μόλις τώρα θα αρχίσουμε την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 7 και θα αρχίσουμε τις ε, προπαρασκευαστικές εργασίες για το 8. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο να μπορέσουμε κατόπιν να βασίσουμε την υπόλοιπη εργασία μας. Υπάρχουν σήμερα τρία βασικά θέματα που θα ήθελα να σας αναπτύξω. Πρώτον, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο, να επιστήσω την προσοχή σας στην υφιστάμενη θεμελίωση της ομάδας εργασίας Ήτρε για την εφαρμογή του πρόγραμματος πλαισίου 7. Και τρίτον, θα κάνω προτάσεις που νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να απλουστευτεί η εφαρμογή των προγραμμάτων έρευνας. Η έκθεση της Επιτροπής Πρώτα, εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το θέμα των ε, γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα. Είναι σοβαρό και δημιουργικό το σχέδιο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η έκθεση της Επιτροπής είναι καλά οργανωμένη, επιτρέπει ιδίως την καθιέρωση προτεραιοτήτων και αποτελεί μια σταδιακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπάρχουν τρία στάδια της απλοποίησης. Πρώτο, μέσα στα πλαίσια των υφισταμένων κανόνων. Δεύτερο, προσαρμογή των κανόνων υπό το φως του συστήματος που ασύζεται στο κόστος. Και τρίτο, μια ενδεχόμενη μελλοντική απλοποίηση που θα σημάνει και μία σε βάθος εξέταση των κανόνων. Οι βασικές επικρίσεις αναφέρονται σε δύο πτυχές. Την σχέση των προτινόμενων αλλαγών με τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανονισμούς και κανόνες συμμετοχής που δεν είναι σαφείς. Εξηγώ. Ορισμένα από τα μέτρα που ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτούν αλλαγή της δημοσιονομικής προοπτικής. Αλλά δεν απαιτούν αλλαγές στους κανόνες. Δεύτερο, ανησυχίες. Ανησυχώ ιδιαίτερα για την διασύνδεση μεταξύ χρηματοδότησης και αποτελεσμάτων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τους κανόνες χρηματοδότησης. Πάντως οι αλλαγές πρέπει να ε, μελετηθούν σοβαρά λαμβάνοντας υπόψη και το, για τις ενδεχόμενες συνέπειες στην ποιότητα της έρευνας και της καινοτομίας. Με ανησυχεί το γεγονός ότι εκ του αποτελέσματος εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε έρευνα που να είναι πιο εγγύς στις απαιτήσεις της αγοράς που δεν είναι επαρκές γιατί χρειάζεται να ε, ε, ενισχύσουμε και την έρευνα που ε, εξετάζει ε, το μέλλον, που στρέφεται προς το μέλλον. Επίσης, αλλαγές μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων κανόνων. Εγώ υποστηρίζω να δοθούν δάνεια μέσα σε μια πλατφόρμα ε, τεχνολογίας της πληροφορικής με ενιαία εφαρμογή των κανόνων σε όλα τα προγράμματα. Για να βελτιστοποιηθεί η δομή και ο χρονισμός των προτάσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, ε, προτά, κάνει προτάσεις σε δύο στάδια. Απαλύνοντας έτσι το, ελαφρώνοντας έτσι το βάρος της υποβολής πλήρων προτάσεων και γι' αυτό η προσέγγιση αυτή σε δύο στάδια πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Εγώ προτείνω να εξεταστούν οι μελλοντικέ τεχνολογίες, το λεγόμενο open scheme, που μπορεί να είναι μια καλή λύση. Η πρακτική της εξέτασης των τιμών δεν πρέπει να γενικευθεί, διότι σημαίνει ότι οι αρχικές φάσεις της έρευνας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και τα περισσότερα πανεπιστήμια και μικρά ερευνητικά κέντρα είναι μικρές και μεσές επιχειρήσεις και εξαρτώνται από εξωτερικούς πόρους για να μπορούν να ασκήσουν την έρευνα. Επίσης, προσαρμογή των κανόνων μέσα στα παρόντα πλαίσια. Προτείνω την εφαρμογή των συνήθων κανόνων για την επιλεξιμότητα και για το κόστος προσωπικού με την ελεύθερη επιλογή κάθε ενός απολύπτη να μπορεί να χρησιμοποιεί είτε το πραγματικό κόστος προσωπικού ή τη μεθοδολογία του μέσου κόστους προσωπικού. Ε, ελεύθερη επιλογή λοιπόν. Υποστηρίζω την ιδέα να εφαρμοστούν τα ίδια funding rates στην, στον υπολογισμό σε όλα τα συστήματα χρηματοδότησης. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού για τα πανεπιστήμια και για τα ερευνητικά ιδρύματα και για τη βιομηχανία, γιατί το κόστος είναι διαφορετικό ανάμεσα σε αυτούς τους φορείς. Η πρόταση να αφαιρεθεί το, ε, τα επιτόκια για τα ε, χρήματα της για τα, χρηματοδότησης είναι σωστή. Κατά αποκοπήν ποσά για το κόστος προσωπικού, ωστόσο πρέπει να βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση. Η πρόταση της Κομισιόν να αφαιρεθούν οι απαιτήσει για τις χώρες μέλη να υποβάλουν γνωμοδοτήσεις πρέπει να συζητηθεί ακόμη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό οι χώρες μέλη να έχουν την ευκαιρία να έχουν την δυνατότητα ελέγχου. Και τέλος το τρίτο, δηλαδή οι πιο ριζοσπαστικές αλλαγές. Σχολιάζω σύντομα τις τρεις επιλογές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη, ειδικά καταπικοποιεί ποσά ανά project ανάλογα με τα αποτελέσματα που ασφαλώς θα μειώσουν το, κόστος, το κόστος αλλά θα σημάνουν δύσκολες διαπραγματεύσεις Είναι δύσκολο να βασιστούν οι χρηματοδοτήσεις στο βέλτιστο αποτέλεσμα, αν βέλτιστο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει ένα πρόσθετο στοιχείο ανταγωνιστικότητα και αυτό είναι καλό. Αλλά θα είναι χαμηλότερη η χρηματοδότηση και μια άλλη παγίδα της επιλογής αυτής είναι ότι θα οδηγήσει σε project που διεξάγονται από κοινοπραξίες που έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν, να επενδύουν σε σημαντική χρηματοδότηση εκτός από τα καταποκοπήν ποσά. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να αποκλείσει ορισμένα πανεπιστήμια και ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τελευταία επιλογή, η τρίτη, είναι η πιο κατάλληλη και οδηγεί στη μεγαλύτερη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους. Το ίδιο προτείνεται δηλαδή και στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Έρευνας. ο κάθε ε, συμμετέχον θα είναι υπεύθυνο για τι δικέ του πράξει. Ένα ενδεχόμενο μειονέκτημα της επιλογή αυτή είναι ότι οι νέοι φορεί ίσως να το βρουν πιο δύσκολο να εισέλθουν στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτά είχα να πω σε σχέση με την έκθεση της Κομισιόν. Τώρα, επιστώ την προσοχή σας, ε, προσοχή σας στην ομάδα εργασίας της Επιτροπής Ήτρε που έχει ήδη υποβάλει ορισμένε προτάσεις και αυτές βέβαια πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεσή μας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις, θα υποβάλω τις γενικές συστάσεις για την έκθεσή μου. Προτείνω ένα σύστημα βασισμένο σε επιστημονική θεμελίωση με έμφαση στην επιστημονική τεχνική πλευρά και στην ε, λεγόμενη peer review, στην, ε, ε, στον έλεγχο δηλαδή των ισοτήμων. Το Κοινοβούλιο την απαλλαγή του ζήτησε να γίνουν αυτές οι απλουστεύσεις. Τρίτο, είναι απαραίτητο είναι απαραίτητο να συζητηθεί εάν απαιτείται για κάθε κανόνα αλλαγή. Η εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών είναι καλή ιδέα. Η εφαρμογή των κανονισμών, των κανόνων μάλλον, σε όλες τις γενικές διευθύνσεις της, της Κομισιόν, τους διαφόρους οργανισμούς, καθώς και στις κοινοπραξίες μεταξύ, ε, με, τα, GTI. Αυτά θα πρέπει όλα να είναι ομοιόμορφα. Όμως θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστούς κανόνες για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια και άλλα για την βιομηχανία και τρίτο και πλαίσιο για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Η απλούστευση χρειάζεται μια προσέγγιση με ανοχή στον κίνδυνο, αποδοχή των γενικών αρχών λογιστικής, αποδοχή των πιστοποιητικών μεθοδολογίας που προβλέπεται από τις εθνικές αρχές. Βελτίωση της πρόσβασης στα συστήματα με καλύτερα εργαλεία ε, τεχνολογίας πληροφορικής και με τους ίδιους κανόνες για όλους τους project officers στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να διατηρούνται οι ίδιοι project officers σε όλη τη διάρκεια των έργων, των project. Καλύτερος χρονισμός των δημοσιεύσεων. Πρόσβαση στα προγράμματα και ούτω καθεξής. Ολοκληρώνοντας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας θα πρέπει να διαπνέονται από πνεύμα εμπιστοσύνης στην επιστημονική κοινότητα και στην ικανότητά της να παραγάγει καινοτομία. Χρειάζεται μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάληψη κινδύνων και στην αποφύγη κινδύνων. Χρειαζόμαστε μια νέα νοοτροπία στην, στην εκτίμηση του κινδύνου για να προσελκύσουμε και νέους φορείς ώστε να γίνει ελκυστικός τόπος η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ερευνητές. Και αναμένω με ενδιαφέρον τη συμβαλή των συναδέλφων μου. Äh, Σας ευχαριστώ. Ήδη ζητούν ορισμένοι τον λόγο. Η κυρία, η κυρία Κωτιά Κορτίνες. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την συνάδελφό μου. Πρόκειται για μια συνάδελφο η οποία πραγματικά γνωρίζει τον κόσμο της έρευνας, γνωρίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, γνωρίζει και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες ευεργετικές ή και καταστροφικές οποιασδήποτε αλλαγής. Οι Beatles επέφεραν επανάσταση στη μουσική και εμείς τώρα χρειαζόμαστε μια τέτοια επανάσταση. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, γιατί διαφορετικά θα επέλθει η καταστροφή. Νομίζω ότι θα επέλθει μεγάλη ε, σύγχυση κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και η εκχώρηση να γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Πέρα από τις συστάσεις της κυρίας Καρβάλιο για μικρότερα προγράμματα, εμείς, η Κομισιόν δηλαδή, προβάλλει μεγάλα προγράμματα. Οι 20-25 πανεπιστημίων δηλαδή, όπου μιλάμε για 5-6 εκατομμύρια ευρώ και τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Εάν θέλουμε να προβάλλουμε μία ε, αν θέλουμε να υπάρχει πραγματική ε, επίπτωση και συνέπεια, θα πρέπει να προβάλλουμε μικρότερα προγράμματα, χωρίς να υπάρχει μία εσωτερική προγενέστερη διεργασία δεν μπορεί να γίνει τίποτα ως προς την έρευνα και την κατάρτιση. Πρέπει να δούμε πώς έχει και το πρόγραμμα υποτροφιών. Στην Ισπανία είναι ξεχωριστό το πρόγραμμα των ε, υποτροφιών. Επίσης δεν έχουμε την κατάλληλη τεχνική υποδομή. Η ΕΠΑ έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τους γιατρούς. Γιατί οι γιατροί δεν είναι βιολόγοι. Αρχίζεται λοιπόν προγράμματα και κλινικών δοκιμών από τη μία πλευρά και προγράμματα ε, υπέρ των ιατρών. Άρα θα πρέπει να έχουμε μικρότερα και πιο εύκολα διαχειρίσιμα προγράμματα και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τις υποτροφίες. Γιατί διαφορετικά δεν θα καλύψουμε την έρευνα. Κολλήγε Τσουκάκης. Κύριε Τσουκάλας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εμπειρία της κυρίας Καρβάλιο με διαβεβαιώνει ότι θα δούμε σύντομα ε, χρήσιμα πράγματα από τον κόπο της. Ε, όμως κύριε Πρόεδρε πρέπει να πω στη σύντομη παρέμβασή μου ότι είμαι απελπισμένος ε, σχετικά με τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν να συμβιβάσουν την απλότητα, την απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης κοινωνικής ε, ευθύνης καθώς και επίσης των αρχών της ε, αριστείας του εξυγχρονισμού του συστήματος κρίσεως από τους ισοτήμους καθώς επίσης και την σημαντική διάσταση ανάμεσα σε αυτό που οι Ευρωπαίοι νομίζουμε ότι είμαστε και σε αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε. Και αυτό που είμαστε είναι ότι δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε τουλάχιστον δεύτεροι. Και ότι οι προοπτικές μας να γίνουμε πρώτοι δεν είναι καλές. Νομίζω ότι αυτές οι σκέψεις και εδώ σταματώ θα έπρεπε να μας οδηγήσουν σε πολύ πιο αποφασιστικές κινήσεις απλούστευσης διαδικασιών όχι σε ένα απείρως πολυπαραμετρικό σύστημα, αλλά με τρεις, τέσσερις, πέντε αρχές που θα στοχεύουν ποσοτικά και ποιοτικά σε αυτά που έχουμε υπόψη μας ότι μας έρχονται ή μας ήρθαν και πάντως όχι αργότερα από το 2020. Η Επιτροπή αυτή κρατάει το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια της. Εάν δείτε μόνο το θεματολόγιο, το σημερινό από Internet Governance μέχρι Pilar de Castillo ε, New Digital Agenda μέχρι Unification of Telecoms και ούτω καθεξής αυτή είναι και η ατζέντα της Ευρώπης από εκεί θα επιβιώσουμε γι' αυτό κάνω έκκληση στην κυρία Καρβάλιο ευχαρίστω θα συνεργαστώ μαζί της για ένα κείμενο που θα κάνει το ΜΕΣ ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο για την εξαιρετική της εργασία επί του δύσκολου αυτού θέματος, διότι εδώ και μερικά χρόνια, 2007-2008, βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες ερευνών μας έχουν επισύρει την προσοχή επί αυτού του θέματος, ότι δηλαδή ε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα ερευνητικά κέντρα, τα κέντρα ερευνών. Η Επιτροπή μας προβάλλει προτάσεις απλούστευσης, χαίρομαι γι' αυτό και την ευχαριστώ για το διάβημα αυτό. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε μια καλή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και να απλουστεύσουμε και τα διαδικαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μας απαντήσει η γραμματεία, αλλά θα, θα έχουμε τελειώσει με τις εκθέσεις πρωτοβουλία. πώς μπορούμε στο δημοσιονομικό κανονισμό να ενσωματώσουμε τις θέσεις μας τη στιγμή που θα γίνει μεταρρύθμιση από την Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολεσμού. Φοβάμαι ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός, μάλλον η αναθεώρησή του, θα έχει κλείσει πριν εγκριθεί η έκθεση πρωτοβουλίας μας. Πώς θα συμφιλιώσουμε το δικό μας λοιπόν χρονοδιάγραμμα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού πρέπει να γνωμοδοτήσει Δεν θα θέλαμε να συμβεί αυτό που συνέβη χθε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των δύο επιτροπών για να έχουμε ένα πολιτικό ε, μήνυμα το οποίο να είναι σαφές. Επί της ουσίας θα εξετάσω ορισμένες προτάσεις από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού όπου συμμετέχω. Θα ήθελα να επισύρω όμως το την προσοχή της εισηγήτριας στην απάτη, σε θέματα απάτης, διότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής γίνεται λόγος για δημοσιονομικούς ελέγχους και για καταπολέμηση της απάτης. Υπάρχει διαφορά μεταξύ σφαλμάτων και απάτης. Διαπράττονται σφάλματα, τα σφάλματα σχετίζονται με την περιπλοκότητα των κανονισμών Απλουστεύοντας τους κανονισμούς θα μειώσουμε και τα λάθη, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την απάτη. Η απάτη είναι ε, κάτι το σκόπιμο, άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Λυπάμαι διότι στο έγγραφο της Επιτροπής υπάρχει σύγχυση ως προς τα σφάλματα και την απάτη. Η Όλαφ έλαβε πολύ αυστηρές ε, αποφάσεις κατά ερευνητών που διέπραξαν σφάλματα. Αλλά ήταν σφάλματα, δεν ήταν σκόπιμη απάτη. Και δυστυχώς κινήθηκε δια της ποινική οδού. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Υπάρχει ένα περιθώριο λάθους, 2%. Θα πρέπει να υπάρχει ανέχεια ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει ανέχεια ως προς τα σφάλματα, αλλά μην γίνεται σύγχυση μεταξύ σφαλμάτων και απάτης. Τι θα κάνουμε με τις προγενέστερες καταστάσεις, διότι υπάρχουν πολλά εκρεμή ζητήματα και νομίζω ότι στην έκθεσή μας θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση έτσι ώστε να κλείσουν όλες οι εκρεμείς διαφορές χωρίς να βρεθούμε ενώπιον δικαστηρίων. Ίσως θα πρέπει να γίνει ένας ε, αντιέλεγχος ή μεταέλεγχος έτσι ώστε να μην γελιοποιηθούμε ενώπιον του ΔΕΚ. Παλτσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την εργασία της και για τις σκέψεις που μας παρουσίασε εδώ σήμερα. Δεν σας λέω τίποτα το καινούριο, θα σας πω ότι ο νέος ευρωπαϊκός ερευνικός χώρος δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί όπως το είχαμε φανταστεί. Ορισμένοι συνάδελφοι πριν από αρκετά χρόνια συζήτησαν ήδη το θέμα, αλλά εμείς ως νέοι ευρωβουλευτές είμαστε κατά κάποιο τρόπο επίσης εμπειρογνώμενες, γιατί στις πατρίδες μας είμαστε σε επαφή με τους ερευνητές. Γι' αυτό οι σκέψεις για την απλούστευση των διαδικασιών και την λύση των ισιών των προβλημάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Από τη σχετική απόφαση θα εξαρτηθεί και η μελλοντική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διέξοδος μας από τη σημερινή οικονομική και νομισματική κρίση. η έρευνα και η καινοτομία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια σχετική καθυστέρηση με άλλες χώρες και αυτό μπορούσαμε να το δούμε και βάσει συγκεκριμένων αριθμητικών στοιχείων. Όπως ανέφερε ήδη η συγγήτρια, χρειαζόμαστε σε ορισμένους τομείς μεταρρυθμίσεις. και θα πρέπει να προτείνουμε λύσεις οι οποίες είναι διαφανείς και θα μας επιτρέπουν τον έλεγχο της χρηματοδότησης. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε απόλυτα αποδεκτές τις προτάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα σχέδια υποδομής στα κράτη-μέλη, γιατί η χρηματοδότηση των μεγάλων ε, έργων υποδομής ε, γίνεται στις παλιές χώρες μέλη και γι' αυτό οι καινούριε χώρες μέλη δεν μπορούν να προχωρήσουν όπως θα έπρεπε στην έρευνα. Θα πρέπει να μελετήσουμε το θέμα, να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Ένα άλλο θέμα είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους επιστήμονες και τους ερευνητές από όλες τις χώρες μέλη. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλό να πετύχουμε επίσης μια ισορροπία μεταξύ της αίτησης αφενός και της ε, πληρωμής της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. <coughs> Καταρχήν, όχι μόνο για λόγου ε, ευγενία, αλλά γενικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, γιατί ο τρόπο με τον οποίο διάστρωσε το θέμα ήταν θαυμάσιο και καλύπτει πραγματικά όλε τι πτυχέ. Ο κύριο Οντί έκανε μια συγκεκριμένη παρατηρήση, δηλαδή το θέμα πώ θα συσχετιστεί αυτή η διαδικασία με όλη τη διαδικασία του προπολογισμού. Πραγματικά για πρώτη φορά μέσα στα πλαίσια αυτής της κοινή ε, ε, ομάδας ψηφοφορία έχουμε τη δυνατότητα αυτή της συνεργασίας. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να μην ακολουθήσουμε μόνο την τόσο ευφυή προσέγγιση της κυρίας Καρβάλιο, αλλά να συσχετίσουμε και με την δημοσιονομική διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βέβαια συζητάμε πολύ το θέμα της, ε, των ποιοτικών προβλημάτων και των ποσοτικών προβλημάτων, αλλά στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα του ποιος είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην έχουμε μόνο ποιοτικές και μόνο ποσοτικές, ε, ποσοτικούς στόχους, αλλά να δούμε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Η απλούστευτη δηλαδή θα πρέπει να έχει και κάποιο benchmark, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μία ε, προσπάθεια για την μείωση της διάρκειας της διαδικασίας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένας ποσοτικός αν θέλετε στόχος. Γιατί αλλιώς την επόμενη ανταθεώρηση δεν θα ξέρουμε τι εξετάζουμε ακριβώς όσον αφορά την απλούστευση. Μια σημαντική ιδέα είναι η αναφορά στις ΜΜΕ. Θα πρέπει εδώ να δούμε ε, ρεαλιστικά ότι η έρευνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προσφανώς πολύ πιο έντονα προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Και αυτό θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο στην απλούστευση να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι σημαντικό αυτό που είπε η εισηγήτρια, ότι θα πρέπει ιδίω για τις ΜΜΕ να έχουμε μία ε, διαφορετική προσέγγιση, γιατί έχουμε αριθμητικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Έχουμε δηλαδή σε διεθνή σύγκριση χαμηλότερη συμμετοχή των ΜΜΕ και επίσης βλέπουμε ότι δεν είμαστε συμφωνοί με την πραγματικότητα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Να έχει δηλαδή διάρκεια αποτελεσμάτων ή μάλλον απόσταση από το αποτέλεσμα από πάνω από ένα χρόνο. Δεν μπορεί να ερευνά απλώς έτσι για την έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μελετήσουμε μήπως θα έπρεπε και εδώ κάπως να τονίσουμε τον στόχο καλύτερα, δηλαδή τη μείωση του χρόνου μεταξύ της αίτησης και της έγκρισης αυτής. Πάντως επαναλαμβάνω ότι η έκθεση ήταν πάρα πολύ ωραία διορθωμένη και θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά γιατί μου φαίνεται ότι η εισηγήτρια πολύ ευφυώς και συναδελφικά έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της κοινή μας ομάδας εργασίας. Και βρισκόμαστε διαφορετικά και όχι εκεί που βρισκόμαστε στην αρχή του 7ου προγράμματος πλαισίου. Πρόεδρος, ναι, σας ευχαριστώ και για αυτό που είπατε, γιατί ήταν μια προσπάθεια που κάναμε, δεν ξέραμε αν θα είχε αποτέλεσμα αυτή η μικρή εργασία που προεργάστηκε. Ο συνάδελφος Ματίας έχει το λόγο. Καταρχήν, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκράσα Καρβάλιο για την εξαιρετική αυτή εργασία. Νομίζω ότι συνοψίζει πολύ καλά την κατάσταση ως προς την πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω ότι εστίασε την προσοχή στα βασικά, στα βασικά σημεία. Θα ήθελα μόνο να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα. Θα έχουμε πολύ καιρό για να εμβαθύνουμε τις συζητήσεις, αλλά θα ήθελα να τονίσω μία από τις μεγάλες μου ανησυχίες. Ξέρουμε ότι είναι πολύ επίγον το ζήτημα. Όλοι μας έχουμε διανύσει μία ε, ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και ξέρουμε ότι τα θέματα απλούστευσης είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία και πώς θα μεταβούμε από το ένα σύστημα χρηματοδότησης στο άλλο δηλαδή ένα σύστημα χρηματοδότησης που να βασίζεται στα αποτελέσματα όπως θέλουμε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που με απασχολούν αλλά και θα ήθελα να το τονίσω διότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να σταθμίσουμε την κατάσταση και να ε, περικλείουμε και ένα σύστημα στάθμισης αποτελεσμάτων. Δεν πρόκειται για μία τόσο ε, απλή διαδικασία αυτή η μετάβαση. Αν θέλουμε δηλαδή να βασιστούμε όχι στο κόστος αλλά στα αποτελέσματα. Πώς θα είναι καλή αυτή η μετάβαση. Εάν λάβουμε υπόψη και το συγκεντρωτικό χαρακτήρα των ερευνητικών κέντρων θα πρέπει να υπάρξουν διαφοροποίησεις και το σημείο κίνησης είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να εμβαθύνουμε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να γίνει απλούστευση, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι τα αποτελέσματα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ανισότητες στο ευρωπαϊκό σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει σύνοχη και να μην ενισχύσουμε τις ανισότητες. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες μου ανησυχίες ως προς την πρόταση της Επιτροπής. Επίσης, Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τα μεγάλα δίκτυα. Η Κομισιόν δεν εμπνέει μία κατάσταση γενικότερης σύνοχης. Θα πρέπει, να δούμε ποιος, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε γιατί νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανισορροπία ως προς την πρόκληση της καινοτομίας. Νομίζω ότι η έρευνα θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των ανησυχιών μας. Είναι μια κινητήρια δύναμη που ορίζει ένα συνεκτικό σύστημα. Όλα αυτά σχετίζονται με την ιστορία μας, με το παρελθόν μας. Νομίζω ότι βεβαίως θα πρέπει να αρκεστούμε στις δυνάμεις μας και ως προς το θέμα της καινοτομίας. Εμείς επενδύσαμε πολύ και χρόνο και δυνάμεις στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε το σύστημα κατά την αλλαγή του. Και ελπίζω να ακουστεί η φωνή μας καθόλου αυτή τη διεργασία και τη διαδικασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκράσα Καρβάλιο για άλλη μια φορά γιατί εργάστηκε πολύ σκληρά για την απλούστευση του συστήματος. Ευχαριστώ, Δικάμπος. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ τη συνάδελφο Γκράσα Καρβάλιο για τον τρόπο παρουσίασης αυτής της έκθεσης και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόν διότι προσπάθησε να αντιμετωπίσει με θάρρος τα προβλήματα και με βάση σκόπιμους μηχανισμούς. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ένα σύστημα αξιολόγησης που προϋπάρχει. Γιατί ήταν ένα καθαρά λογιστικό σύστημα, ενώ τώρα θα πρέπει να έχουμε ε, εταιρικές σχέσεις που να βασίζονται στην εμπιστοσύνη trust-based. Έτσι θα πρέπει να έχουν οι αξιολογήσεις μας. Για πολλά χρόνια οι αξιολογήσεις επιστημονικών προγραμμάτων βασίζονταν στις εργασίες συμβούλων Δηλαδή έβρισκαν μία αναλογική σχέση η οποία όμως στην ουσία δεν υπήρχε. Εδώ μιλάμε για επιστημονικές διεργασίες. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μία ισορροπία που δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει να χωρίσουμε τα project σε μεγαλύτερα και μικρότερα. Μεγαλύτερης και μικρότερης εμβέλειας. Έτσι ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς έχει γεωγραφική κατανομή των ε, προτάσεων. Γι' αυτό και οι κοινοπραξίες είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλίσουμε αυτή τη γεωγραφική διαφοροποίηση. Επίσης, θα πρέπει να μιλάμε για βασική έρευνα και καινοτομία. Δεν θα πρέπει να ζητάμε υπερβολική καινοτομία και όπως είπε η Μαρίζα Ματίας να εγκαταλείψουμε τη βασική έρευνα. Θα πρέπει να βασιστούμε στην πείρα μας. Υπάρχει το European Research Council, στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε. Δηλαδή βασιζόμαστε σε ε, μεθόδους αριστείας. Αλλά δεν είναι ε, μοναδική αυτή η μέθοδος γιατί έτσι μπορεί να επέλθει γεωγραφικός συγκεντρωτισμός ως προς τις υποψηφιότητες. Ένα από τα πιο δελεαστικά στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Καρβάλιο είναι τα, η παρουσίαση των υπέρ και, τα, και των κατά. Θα πρέπει να επέλθει μια σωστή ισορροπία στην κατανομή και την επιλογή. Θα πρέπει να ζητήσουμε απλούστευση, αλλά οπωσδήποτε τα tailor-made προγράμματα δεν είναι τα καλύτερα Δυστυχώς η γραφειοκρατία πάντα υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς ως προς την αξιολόγηση. Αυτή την οδό νομίζω ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Uh, important uh, file, uh, but it Σημαντικό αλλά δύσκολο θέμα. Αφενός πρέπει να απλουστεύσουμε, αλλιώς οι μικρές επιχειρήσεις θα κάνουν και λιγότερη έρευνα και, τα μικρά επιστημονικά ιδρύματα το έχουν πάρει απόφαση νομίζω πια ότι θα συμμετέχουν όλο και λιγότερο σε ερευνητικά προγράμματα. Από την άλλη μεριά οφείλουμε να διατηρήσουμε κάποιο έλεγχο. Οι θέσεις μας ως πρασίνων είναι ότι πρέπει να επιφέρουμε κάποια διαφορά, να υπάρχει κάποια διαφορά δηλαδή. Εάν πρόκειται για project κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό πρέπει να πετύχουμε εδώ. Δεν εκπλήσωμε από την ποιότητα της εργασίας της εισηγητρίας, η οποία είναι την ποιοτητα της εργασιας της συγκεντριας γνώστης του θέματος. γενικά θα ακολουθήσουμε τη γραμμή της. Σας ευχαριστώ κύριε Τούρμες. Del Castillo. Ε, mm, θα επαναλάβω αυτά που προείπαν και άλλοι. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, διότι ε, επετέλεσε ένα εξαιρετικό έργο, πολύ καλά διαρθρωμένο κάτι το οποίο είναι πραγματικά ε, ε, επενεταίο. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά που είπε ο κύριος Οντί είναι πολύ σωστά σε σχέση με τις δημοσιονομικές ανάγκες και να τονίσω το εξής. Μέχρι το μέσον της θητείας ο τομέας της έρευνας θα είναι το επίκεντρό μας, διότι βεβαίως έχει οριζόντιο χαρακτήρα και σχετίζεται και με άλλους τομείς. Δηλαδή με έργο άλλων επιτροπών. Θα πρέπει όμως να ε, πρόκειται για μια συνεκτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα λάβουμε μια απόφαση μεγάλης εμβέλειας που είναι το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο θα προταθεί από την ε, Κομισιόν στις αρχές του επόμενου έτους, αλλά έχουμε την πρώτη αυτή έκθεση για την ε, απλοποίηση, για την απλούστευση. Έχουμε την ε, ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Έχουμε τους διαδικαστικούς κανόνες, το πρόγραμμα πλαίσιο και τις πέντε εκθέσεις νομοθετικού περιεχομένου που συνδέονται με το πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ε, μεγάλο εκτενές πακέτο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου την κατάσταση κρίσης στην οποία βρισκόμαστε και διανύουμε. Νομίζω λοιπόν ότι με βάση τη μικρή μας ε, μέχρι τούδε πείρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά που μας προτείνει η κυρία Καρβάλιο γιατί θα ασχοληθούμε όχι μόνο εμείς που είμαστε σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και άλλοι. Θα πρέπει η επιτροπή αυτή να είναι μία μόνιμη επιτροπή. Μέχρι ότου λήξουν όλα τα θέματα απλούστευσης. Στο, δηλαδή μέχρι την έγκριση του 8ου προγράμματος πλαισίου. Και τα συμπεράσματα της ε, Επιτροπής να γνωστοποιηθούν. Δηλαδή, σε τακτά χρονικά διαστήματα να αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της ε, Ήτρε μία ανακεφαλαίωση των ε, εργασιών. Δεν χρειάζονται μεγάλες ε, συνεδριάσεις. Θα πρέπει η Επιτροπή αυτή να μας μιλά για τα συμπεράσματά της. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα στον τομέα των απλουστεύσεων. Και αυτή η ανακεφαλαίωση να αποσταλεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Άρα, από πλευράς εσωτερικών διαδικασιών, αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι ένα θέμα προτεραιοτήτων. Έτσι ώστε το έγγραφο αυτό να το έχουμε όλοι στη διαθέσή μας. Θα διανεμηθεί και το έγγραφο. Ακόμη δύο, αλλά πρέπει να βιαστούμε λίγο. Βανίστε Ρόι. Ευχαριστώ. Κάτι σχετικό με τις διαδικασίες, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που είπαν άλλοι πριν. Έχουμε πολλές ιδέες σχετικά με την απλοποίηση και γνωρίζουμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην πράξη. Αυτό που νομίζω ότι λείπει εδώ είναι ότι βλέπουμε ε, εγκαίρως κάποια σημεία Βλέπουμε για παράδειγμα τις ε, κοινοπραξίες ε, τεχνολογικής καινοτομίας όπου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραγωνίζονται. Τα χρήματα που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα φαίνεται τελικά να μην καταλήγουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα πάρουμε κάποια απόφαση τώρα ή θα τα αναβάλουμε όλα για το 2013 τα διαρθωτικά ταμεία, το περιφερειακό ταμείο πρέπει να επανεξεταστούν. Χρειάστηκε να επανεξεταστούν μάλιστα δύο φορές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις τώρα και όχι να περιμένουμε. Κάποιος είπε πριν ότι θα τα κάνουμε αυτά το 2013. Αυτό είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η πρόταση για αναθεώρηση μετά τριετία της δημοσιονομικής προοπτικής βασίζεται ωστόσο, άπτεται μάλλον των βασικών αρχών που πρέπει να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε αφενός την παρούσα προσέγγιση όπως είπε και η κυρία Καρβάγιο. Δεύτερο θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια ξεκάθαρα σημάδια σχετικά με την δημοσιονομική προοπτική Όλη η συζήτηση που γίνεται γύρω από την ε, υπερβολική γραφειοκρατία, τον περισσότερο έλεγχο κλπ. Αυτά αρχίζουν και κυριαρχούν εδώ, ενώ εμείς θέλουμε να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Δεν θέλουμε να ρίξουμε υπερβολικό βάρος στην τήρηση και του τελευταίου γράμματος. Έχω όμως και άλλο ένα σχόλιο. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Χατζημαρκάκη, μιλήσαμε πριν μαζί του έχουμε πρόσθετα πρόσθετους πόρους, έχουμε και κάποιες συστάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί περισσότερη συνέργεια. Άλλωστε ψηφίστηκε κάτι σχετικό στην Ολομέλεια και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό, δηλαδή να βελτιωθεί η λεγόμενη στα αγγλικά synergy, εν πάση περιπτώσει. Εμείς πληρώνουμε το 5% του προϋπολογισμού εγώ νομίζω ότι χρειάζεται καλύτερη διασύνδεση μεταξύ του δικού μας προπολογισμού, των κριτηρίων, των προτεραιοτήτων και την μείωση τη γραφειοκρατίας. Ακούμε συχνά ότι θα είναι σημαντικά τα ωφέλη εάν το επιτύχουμε. Καλά, θα αρκεστώ σε αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία. Ο κ. Χατζημαρκάκης. Έπαινος και στην Κομισιόν και στην εισηγήτρια. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι σημαντικό αλλά είναι και δύσκολο. Έχουμε μπροστά μας μια κατάσταση όπου οι πόροι σπανίζουν όλο και περισσότερο. Τα χρήματα θα λείπουν όλο και περισσότερο. Αν επιτρέψουμε τώρα να υπάρχει μια πολιτική ε, πρόθεση της έρευνας χωρίς συνοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι πλέον αποδεκτή η κατάσταση αυτή. Και γι' αυτό χαίρομαι που έγκαιρα τώρα, πριν από το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, συζητούμε το θέμα αυτό. Και ο κ. Σόντι και εγώ είμαστε και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και γνωρίζουμε ότι ευθύνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αύξηση της γραφειοκρατίας. Και γι' αυτό χρειάζεται τώρα να σφίξουμε λίγο τα λουριά. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προτάσεις. Αν προτάσεις είναι καλές. Δεν είναι όμως μόνο οι πόροι. Γίνονται όλο και πιο αόρατα τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα. Ποια είναι τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που αν βγει κάποιο και μα ρωτήσει, μα τι κάνετε στην Ευρώπη, να ξέρουμε να δώσουμε μια απάντηση αμέσω. Ωραία, το ITER, το Airbus και τελείωσε. Δεν υπάρχουν τα μεγάλα αυτά ερευνητικά προγράμματα που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι ορατά τα προγράμματα αυτά. Και μπαίνει και ένας τρίτος προβληματισμός. Η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Έρευνας η οποία αμφισβητείται όλο και περισσότερο. Έχουμε από τις εκλογικέ μας περιφέρειες ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στα γραφεία μας και μας λένε αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν μας ωφελούν. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν, να ταρκουνηθεί το σύστημα. Όπως είπε ο Βανίστελ Ροϊ πριν, αγωνιζόμαστε ώστε όχι μόνο στον τομέα πρόθεση της έρευνας, αλλά και σε όλους τους άλλους, περιφερειακό, ενίσχυση των διαστατικών ταμείων και το να υπάρξουν οι ίδιες συνθήκες για την υποβολή των αιτήσεων. Αυτά είναι δυνατόν να γίνουν, διότι εν τέλει τεχνικά προβλήματα. Αυτά λοιπόν που προτάθηκαν, δηλαδή να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αυτά είναι τεχνικά ναι, αλλά και πολιτικώς εφικτά. Το τρίτο ε, σύνολο θεμάτων είναι πολιτικά δυσκολότερο. Δηλαδή, να γίνει επιστημονικά θεμελιωμένη ε, έρευνα η οποία να κρίνεται εκ του αποτελέσματος και αυτό είναι νέο στοιχείο. Και γι' αυτό άκουσα και αυτά που είπαν οι Πορτογάλοι συνάδελφοι οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ε, βασικής έρευνας αλλά έχουμε και ένα παράδειγμα όπου το Συμβούλιο Έρευνας δίνει κατά αποκοπήν ποσά ένα είδος επιβράβευσης όταν επιτυγχάνονται κάποια αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Συμβούλιο Έρευνας δείχνει ότι είναι δυνατόν και στην έρευνα βάσης να γίνει, να εφαρμοστεί αυτό. Ας ε, αποφασίσουμε λοιπόν και εμείς να ε, ενισχύσουμε αυτή την έρευνα βάσης κρινόμενοι και εκ του αποτελέσματο. Χρειαζόμαστε αλλαγή παραδειγμάτων στην πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε μια πρώιμη φάση. Α εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μα δίνεται. Είδε μη, ο κόσμο θα μα γυρίσει την πλάτη. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι όλο και λιγότερου θα έχουμε που θα ζητούν χρηματοδοτήσει, κυρίω από τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Παρακαλώ να προχωρήσουμε λίγο σύντομα. Σάρος. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό που συζητούμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια και νομίζω ότι πρέπει όντως να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Εξετάζοντας την διοικητική πλευρά των ερευνητικών προγραμμάτων και εγώ έχω γνώση γιατί ήμουν και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ περίπλοκα. Πολλοί ερευνητές έχουν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα. Άλλοι όμως αρνήθηκαν διότι θεώρησαν ότι ήταν υπερβολική η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Έχω λοιπόν να πω το εξή. Η απλοποίηση μπορεί να αποτελέσει για μας ένα εργαλείο, ένα μέσον για να ενισχύσουμε ορισμένους τομείς της έρευνας. κάνοντας και τη χρηματοδότηση λοιπόν πολύ ελκυστικότερη για τους ε, ερευνητές και αναφέρομαι σε τομείς όπως της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας, των ε, κλιματικών αλλαγών και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να περιληφθούν σε αυτή τη μελλοντική προσπάθεια. Εκ. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση. Υπενθυμίζω ότι ήταν ανησυχητικά τα συμπεράσματα της μήνυ ακρόασης που κάναμε το προηγούμενο φθινόπωρο εδώ στην Επιτροπή μας για την μείωση της γραφειοκρατίας. Με την εξαιρετική εισηγήτρια κυρία Καρβάιο είμαι βέβαια ότι θα περιληφθούν τα συμπεράσματα της ακρόασης αυτής στην έκθεση. Έγινε και μια στρογγυλή τράπεζα στην Ισπανική Προεδρία με πολύ εξαιρετικά συμπεράσματα που πρέπει επίσης να σημειώσουμε. Εν τέλει, ο συνδυασμός των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων, του προπολογισμού δηλαδή, και των πρόσφατων συζητήσεων που διεξαγάγαμε. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Οι διάφορε πολιτικές ομάδες να εξετάσουν τις διάφορε γραμμές του προπολογισμού. Διότι εξετάζοντας τα κονδύλια αυτά θα δούμε ότι άπτονται ορισμένων από τι προτεραιότητε τη επιτροπή μα, Άρα χρειάζεται συνδυασμό των συζητήσεων που έχουμε κάνει για την έρευνα με, τον, με τις συζητήσεις που κάνουμε για τον προπολογισμό. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική συζήτηση. Έγινε και η προσπάθεια να γίνει μια καινούργια αφετηρία με τη μικρή αυτή ομάδα εργασία. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι βεβαίω σήμερα παρούσα ότι δεν θα μπορέσουμε να τη δώσουμε, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη δώσουμε σήμερα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εδώ λίγη η συνεδρίαση και ευθύ αμέσω θα παρακαλέσω να εγκαταλείψουν την αίθουσα οι συνάδελφοί μας που δεν είναι συντονιστές και να παραμείνουν συντονιστές.